Chers collègues, bonjour à tous. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ας περάσουμε σύντομα στην έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Φαντάζομαι δεν προτείνονται αλλαγές, άρα μπορούμε να την εγκρίνουμε. Και να περάσω αμέσως στο σημείο 2 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει δύναμη το άρθρο 118 στα πλαίσια της ε, προετοιμασίας ε, της επανεξέτασης για το 2020 της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών μία σύσταση στην του, ε, στον ύπατη εκπρόσωπο του Συμβουλίου για τον έλεγχο και την, τον πυρηνικό εφοπλισμό. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε στις 23 Ιανουαρίου στην ΥΠΑ και η έγκριση στην ε, Ολομέλεια θα γίνει στην εβδομάδα 14, τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου, Μαρτίου δηλαδή. Επίσης αποφασίσαμε να εγκρίνουμε έκθεση πρωτοβουλία για τις προκλήσεις και προοπτικές των πολυμερών συστημάτων ελέγχου όπλων και αφοπλισμού με εισηγητή τον κύριο Σβέν Μίξερ. Η πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της δέκατης διάσκεψης επανεξέτασης της συνθήκης περιμηδιάδοση κάτι που είναι συνετό κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Ιζούμι Νακάμιτσου, βοηθό του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είπα ότι εκπρόσωπο για θέματα αφοπλισμού. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω θερμά που δέχτηκε την πρόσκλησή μα να λάβει μέρο σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη τη Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα. Ε, και τα μέλη τη αντιπροσωπη για τη σχέση με τι ηνωμενε πολιτειε Μάλιστα καλωσορίζω την κυρία τζακι Τζόου, την πρόεδρο τη αντιπροσωπη αυτη Συναντηθήκαμε στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019 στα πλαίσια μια αποστολή υποεπιτροπή μα στα Ηνωμένα Έθνη και σήμερα ξαναβρισκόμαστε εδώ στη στι εγκαταστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι Βρυξέλλε, για να αγγίψουμε σε ένα θέμα που απέκτησε κρίσιμο χαρακτήρα τον τελευταίο καιρό, την διαδικασία επανεξέταση το 2020 τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών και το μέλλον του ελέγχου των πυρηνικών όπλων και του πυρηνικού αφοπλισμού. Μάλιστα, εορτάζουμε φέτο την 50η επέτειο τη συνθήκη περί διάδοση, που είναι ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου συστήματο αφοπλισμού και μη διάδοση των πυρηνικών. Και μάλιστα από τη θέση ισχύ του 70, η συνθήκη αυτή συνέβαλε στη μείωση τη διάδοση των πυρηνικών και στη μείωση του πυρηνικού προστασίου. διευκόλυνε την ειρηνική χρήση τη πυρηνική ενέργεια και δημιούργησε, ε, ευνόησε μάλλον τη δημιουργία ζωνών χωρίς πυρηνικά. Στα, πλέξια, στα σημερινά πλαίσια της ε, ταχύτητα της επιδείνωσης της ε, διεθνούς ασφάλειας, ο ρόλος και η σημασία των πυρηνικών ε, βρίσκονται πλέον στη διεθνή προσοχή. Και η αυξανόμενη καχυποψία μεταξύ των κρατών και ο εξυγχρονισμό των αποστασίων λόγω των νέων τεχνολογιών είναι υποκείμενε αιτίε. Οι κίνδυνοι μάλιστα για την ασφάλεια έχουν οξυνθεί από πιθανές επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις στα πυρηνικά όπλα και στα συστήματα δίκης και ελέγχου τους. Σε λίγους μήνες θα, θα περάσουμε στην δέκατη διαδικασία επανεξέτασης της ήθικης διάδοσης Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ δύσκολες ε, λόγω της έλλειψης ε, πρόοδου στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, την αποχώρηση των ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση και από τι ε, μόνιμες παραβάσει ε, τη πυρηνικής συμφωνία από το Ιράν, κάτι που ενεργοποίησε το μηχανισμό επίλυση των διαφορών από τη Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε η συζήτηση δεδομένης και της τελευταίας έλλειψης ε, πρόοδου του 2015 ε, οι διαπραγματεύσεις προμηνύονται δύσκολες. Βέβαια, στην επερχόμενη διάσκεψη για την επανεξέταση θα πρέπει να σημειώσουμε αυτή την πρόοδο και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη για να βοηθήσουμε τη δημιουργία διαλόγου προκειμένου να καταλήξουμε σε αποτελέσματα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη βρίσκοντα τα κοινά σημεία των διαπραγματεύσεων. Είναι προς όφελος όλων μας να διαφυλάξουμε αυτή την παγκόσμια αρχιτεκτονική αφοπλισμού. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνθήκη και τους ε, τρεις πυλώνες της ε, που χαρακτηρίζονται από ελεξάρτηση και αλληλοσυμπλήρωση. Θα πρέπει επίσης να υλοποιήσουμε τα διαδοχικά στάδια προκειμένου να καταλήξουμε σε πυρηνικό αφοπλισμό και να μειώσουμε τη σημασία των πυρηνικών όπλων στι εθνικές πολιτικές και δόγματα, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να μειώσουμε τον πυρηνικό κίνδυνο και να καθιερώσουμε τη μη χρήση των πυρηνικών ως υποχρεωτικού και απαράβατου κανόνα. Και μάλιστα πρόσφατα το πέρυσι η κατάρρευση μιας άλλη σημαντική συμφωνία, τη συνθήκη για τα πυρηνικά μέσου βεληνικού, που για δεκαετίε ήταν ακρογωνιαίος λίθος της ε, παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, απίθυνε επίγουσα έκκληση προς τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για να ξεκινήσουν διμερή επικοδομητικό διάλογο και να έχουν διαπραγματεύσει και με άλλα κρατημέλη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα θέλαμε οι δύο χώρε να ξαναρχίσουν το διάλογο προκειμένου να καταλήξουν σε ένα δεσμευτικά, νομικά δεσμευτικό ε, μηχανισμό για τους πυράβλους ε, μικρού και μέσου βεληνικούς και να ε, δεσμευτούν και μάλιστα πριν τη διάσκεψη για τη μη διάδοση να παρατείνουν την συνθήκη για τη νέα συμφωνία για μία των στρατηγικών όπλων. Βρισκόμαστε στο παραπέντε πριν διαλυθεί τελείως το Παγκόσμιο Σύστημα Ελέγχου των Όπλων. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένα Έθνη τις προσπάθειες, ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε στη συνθήκη για τη μη διάδοση για την επόμενη δεκαετία. Κύριε Νακαμίτσο, αναγνωρίζουμε ότι το έργο σας δεν είναι το, και το πιο εύκολο, αλλά σας διαβεβαιώνω για την αμέριστη υποστήριξη των μελών της Υποεπιτροπής σε αυτό σας το εγχείρημα. Και θα σας δώσω το λόγο. Thank you so much, Madam Chair, for this, um, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετικά ευγενική αλλά και πολύ ουσιαστική σας ε, εισαγωγή στα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στην ε, κύρια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αφοπλισμό. Θα εστιάσω ιδιαίτερα στην 22η σύμβαση, ε, συνέλευση μάλλον αναθεώρησης του TNP, ε, τις συνθήκες για τη μη διάδοση των πυρηνικών, αλλά θα εστιάσω και στα ζητήματα ε, της, ε, του ελέγχου των στατηγικών όπλων και του αφοπλισμού σε πολλά σημεία του κόσμου. Ε, ακούγονται πολλές επικρίσεις και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και βεβαίως θα μιλήσουμε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτούς τους τομείς. Για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιστεύω πως ο αφοπλισμός είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Στα Ηνωμένα Έθνη συχνά μιλάμε για την επιδείνωση της κατάστασης ε, της διεθνούς ασφάλειας και πιστεύω πως και εσείς ε, το αισθάνεστε σε αυτή την ήπειρο ιδιαίτερο αυτό. Να πω εξ αρχής ότι στον ΟΗΕ ε, βλέπουμε τον έλεγχο όπλων, την μη διάδοση και τον αφοπλισμό ως μέσα ή εργαλεία για την επίτευξη της ασφάλειας. Δεν πρόκειται για οτοπικά όνειρα, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο τον αφεπλισμό, γιατί ακριβώς επιθυμούμε ασφαλέστερο κόσμο. Και από αυτή την άποψη το γεγονός ότι το έλεγχος των όπλων, η διαφάνεια και τα μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θεσπίστηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ψυχρού πολέμου και βεβαίως και μετά Αυτά όλα συνέβησαν γιατί πολλές χώρες ολόκληρο τον κόσμο θεώρησαν ότι τα μέσα αυτά θα ήταν ακριβώς χρήσιμα για την ασφάλεια, ιδιαίτερα σε αυτό το πλαίσιο. Αναφέρατε ήδη, κυρία Πρόεδρε, την συνθήκη INF για τα πυρηνικά μέσου βεληνικούς, ιδιαίτερα όσον στη διάρκεια της κρίσης των ε, πυράβλων και βέβαια ε, ε, θυμίζουμε ότι και πάλι αναμένουμε, μάλλον είμαστε εκτεθειμένοι την απειλή των όπλων ε, μέσου ελληνικού και πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αισθανόμαστε μάλλον τη, την ίδια αίσθηση να επανέρχεται με πιο απρόβλεπτο και ασταθή τρόπο και γι' αυτό θεωρούμε ότι για να προδεύσουμε και να βαθύνουμε τις συζητήσεις για τα θέματα ελέγχου των εξοπλισμών, του αφοπλισμού και της ε, μη εξάπλωση των πυρηνικών είναι ε, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Και ε, Γι' αυτό και το 2020 έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ε, φέρνει διάφορα σημεία επαφής που και προβληματισμού που αποτελούν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους όσον αφορά την παγκόσμια προσπάθεια εφοπλισμού και όπως αναφέρατε ίσως η πιο σημαντική είναι η συνέλευση αναθεώρησης της συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Θα επανέλθω σε λίγο σε αυτήν και θα μιλήσω πιο αναλυτικά αλλά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη έχουν ε, ε, εισακουστεί και θεωρούνται ως οι βασικοί ε, υποστηρικτές της μη εξάπλωσης και του αφοπλισμού. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον ΟΙΕ, ο οποίος από την ίδρυσή του έχει καταβάλει προσπάθειες για να επιτύχει την πλήρη εξάλληψη των πυρηνικών όπλων και των άλλων όπλων μαζικής καταστροφής και γι' αυτό εξ αρχή θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη τη για την υποστήριξη και τη συνεργασία στον ΟΗΕ ώστε να ακούγονται αυτές οι απόψεις που είναι τόσο σημαντικές για μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ελπίζω να το γνωρίζετε, αλλά ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2018 ξεκίνησε την ατζέντα για τον αφοπλισμό ε, για την εξασφάλιση του κοινού μας μέλλοντας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη μάλλον εκτίμηση της κατάστασης και περιλαμβάνει και μια σειρά από πολύ πρακτικές προτάσεις για το πώς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ μπορούν να προωθήσουν τον αφοπλισμό και συμπεριλαμβάνει επίσης 40 πολύ συγκεκριμένες ε, δράσεις. Και πάλι είμαι ευγνώμων γιατί μπορώ να πω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε σταθερά και έχει πρωτοστατήσει σε πολλά από αυτά τα σημεία δράσης και πάντοτε είναι ευχαρίστησή μου για μένα στα Ηνωμένα Έθνη να μπορώ να συνεργάζομαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα. Να ξεκινήσω με την συνέλευση για την αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη 27 Απριλίου με 22 Μαΐου και πρόκειται για μια συνέλευση που θα αφορά την ίδια ε, τη συνθήκη. Πρόκειται για την 50η επέτειο της συνθήκης αυτής, της έναξης και 25η επέτειος της επαόριστον παράτασής της. Η συνθήκη, πιστεύω όλοι θα συμφωνείτε, εξακολουθεί να αποδίδει ε, και να επιφέρει πολύ απτά ε, ωφέλη ως προς την ασφάλεια. Για παράδειγμα, επιβάλλει ε, επαληθεύσιμες υποχρεώσεις ε, στα κράτη που δεν έχουν πυρηνικά όπλα να μην αποκτήσουν και να μην αναπτύξουν δικά τους. Ε, και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της διεθνούς κοινότητας. Επίσης, η συνθήκη αυτή περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές ε, υποχρεώσεις για όλα τα συμβαλόμενα μέρη για την επίτευξη της εξάλληψης των πυρηνικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των μοναδικών υποχρεώσεων που βασίζονται σε συνθήκη που έχουν υπογράψει τα πέντε πυρηνικά κράτη ε, που είναι συμβαλόμενα μέρη. Νομίζω λοιπόν πως είναι πολύ σημαντική αυτή η συνέλευση για την μεταρρύθμιση και, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την επέτειο στον ΟΙΕ. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Να σας αναφέρω τρεις εξ αυτών. Η πρώτη είναι βέβαια η επιδείνωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας που ανέφερα νωρίτερα, πράγμα που θα έχει από, το, από, ε, την, ε, από την επιρροή στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα στα πέντε πυρηνικά κράτη που είναι πηγή ανησυχίας. Μέχρι στιγμής τα πέντε πυρηνικά κράτη ανέκαθεν μοιράζονταν πολύ ε, έντονα συμφέροντα ώστε να εξασφαλίσουν πως η συνθήκη θα ε, παραμείνει υγιής και ισχυρή, όμως έχει παρατηρηθεί ότι η συμφωνία μεταξύ των πέντε αυτών συμβαλωμένων κρατών κάπως αποδυναμώνεται. Θα είναι λοιπόν μια στρατηγική πρόκληση αυτή που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεύτερο ζήτημα είναι οι περιφερειακές διανέξεις που μπορεί να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα και όλος ιδιαίτερος οι συνεχιζόμενες διαφωνίες σε σχέση με ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ξέρω πως αυτό είναι πολύ ε, ανησυχητικό θέμα και για σας, αλλά στο πλαίσιο της συνθήκης επίσης ε, μας προβληματίζει. Τρίτη σημείο είναι βεβαίως η ε, ο προβληματισμός των μη πυρηνικών κρατών μελών σε σχέση με την έλλειψη προόδου προς την, τον πυρηνικό αφοπλισμό σας ανέφερα ότι τα πυρηνικά κράτη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις που είναι νομικά δεσμευτικές μάλιστα ε, όσον αφορά τον αφοπλισμό αλλά έχει υπάρξει πολύ ίχνη πρόοδο τα τελευταία χρόνια ιδίω και αυτό προβληματίζει πολύ τα μη πυρηνικά ε, κράτη. Έχει παρατηρηθεί ότι μία από τις ε, εσωτερικές ε, ε, τους ιστορικούς προγραμματισμούς αφορούσε την ισορροπημένη εφαρμογή της συνθήκης στους τρεις πυλώνες της ε, σημαίνει ειρηνική χρήση, μη εξάπλωση και αφοπλισμό. Υπάρχει έλλειψη προόδου και μάλιστα και αντιστροφή, οπισθοδρόμηση μάλλον των προγραμμάτων. Μιλήσατε, Πρόεδρε, για τον εξυγχρονισμό και όπως καταλαβαίνετε αυτό αμφισβητεί πολύ το αν υπάρχει πρόοδος ή όχι. Και αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ όσον αφορά τις δεσμεύσεις ε, αφοπλισμού που ανελήφθησαν το 2000 και το 2010 στις αντίστοιχες ε, ε, συνελεύσεις. Αυτές είναι οι σοβαρότερες προκλήσεις που παρατηρούμε πριν την συνέλευση του 2020. Τα κράτη-μέλη δαπανούν πολύ χρόνο εξετάζοντας τι σχήμα θα, έχει, θα έχουν τα πορίσματα της συνέλευσης του 2020 και τι ζητήματα θα βρουν αρκετή υποστήριξη ώστε να περιληφθούν εκεί. Έχουν ήδη υπάρξει πολλές διαβουλεύσεις και επίσημες συζητήσεις. Υπάρχουν ζητήματα σαφώς που δεν μπορούν να επιληφθούν πριν τη συνέλευση. Τα κράτη-μέλη θα, θα συγκεντρωθούν. Ε, η συνέλευση θα διαρκέσει ένα μήνα. Οπότε τα θα εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε ήδη κάποια στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν ε, τμήμα οποιοδήποτε τελικού αποτελέσματος. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι θα περιληφθούν στα πορίσματα του Μαΐου φέτος. Το πρώτο, ελπίζω, θα είναι η επαναδιατύπωση των συμπεφωνημένων ε, υποχρεώσεων από προηγούμενες διασκέψεις και επίσης μια νέα πολιτική δέσμευση να επιταχυνθεί η εφαρμογή συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνηση συγκεκριμένων οροσίμων για να μπορούμε να παρακολουθούμε την επίτευξη προέδου, πρόοδου. Δεύτερον, ενισχυμένη πρόσβαση στην ε, ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας και επίσης ε, θέλουμε να προωθήσουμε την ε, εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και η δέσμευση να ενισχυθεί η μη, διάδοση, η και τα μέτρα της μη διάδοσης, κυρίως υπό το φως ε, των πιθανών τροτών σημείων που έχουν αναδειχθεί λόγω των προκλήσεων των νέων τεχνολογιών, όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε. Και τέταρτο, γενική διερεύνηση πρακτικών μέτρων. Σίγουρα το περιβάλλον ασφάλειας ε, είναι αντίξω, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά ε, απτά και συγκεκριμένα για να προωθήσουμε ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά και να κάνουμε κάποια βήματα για να μειώσουμε τον πυρηνικό κίνδυνο και να στηρίξουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ε, των προτύπων επαλήθευσης του πυρηνικού αφοπλισμού. Αυτές είναι ιδιαίτερα τεχνικές συζητήσεις, αλλά είναι εφικτές σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων που θα συζητήσουν τα τεχνικά σημεία και τις ικανότητες ε, που, υπάρχει, που υπάρχουν για την επαλήθευση του πυρηνικού αφοπλισμού. Οπότε αυτές ε, οι προτάσεις και ιδέες ήδη έχουν ανακύψει στην προπαρασκευαστική φάση της επόμενης διάσκεψης. Και μάλιστα ο πρόεδρος της επόμενης διάσκεψης ε, είναι ο πρέσβης Γουστάβος Όλμπινεν, που θα παραβρεθεί αύριο στη Γενέβη και εγώ θα μεταβώ αύριο στη Γενέβη και αδειμονώ να τον συναντήσω για να συζητήσουμε πιο διεξοδικά μερικά από τα θέματα αυτά. Επίσης, ε, θα γίνει μια σημαντική προπαρασκευαστική συζήτηση στη Γενέβη για όλα αυτά τα ζητήματα. Και από ευκαιρία θα ήθελα να πω πόσο ανεκτήμητη ήταν η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία αυτών των συνεδριάσεων και των διαβουλεύσεων, τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Οπότε, σε τελική ανάλυση, ο διάλογο και η αναγνώριση των εύλογων και θεμητών ανησυχιών όλων των συμβαλωμένων κρατών, ιδιαίτερα εν ώψη της επιδείνωση της κατάστασης ασφάλεια παγκοσμίω και ένα πνεύμα ευελιξίας ε, θα χρειαστούν οπωσδήποτε για να ευοδοθεί η διάσκεψη επανεξέτασης. Και από αυτήν την άποψη θα χρειαστεί ηγετικός ρόλος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να συμβάλλουν σημαντικά προκειμένου να δημιουργήσουν γέφυρες, να διευκολύνουν το διάλογο και να ταχθούν υπέρ ενός ε, αισιού αποτελέσματος. Υπάρχει μεγάλη διαφωνία και διάσταση απόψεων μέχρι στιγμής και γι' αυτό προσβλέπουμε στην υποστήριξη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διευκολύνουμε τη συζήτηση και να εισακουστεί η έκκληση για ευελιξία, ελαστικότητα στην προσέγγιση των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων και με ένα συμβαστικό και συνεργάσιμο πνεύμα. Όλα αυτά θα είναι απολύτως απαραίτητα για να τελεσφορήσει η διάσκεψη επανεξέτασης. Και προσβλέπουμε στον επικοδομητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο από τις πέντε πυρηνικές δυνάμεις ε, του TMP και έχει στενές σχέσεις με τις άλλες τρεις πυρηνικές δυνάμεις της συνθήκης περιμηδιάζωσης των πυρηνικών. Οπότε έχουμε πολλά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ του αφοπλισμού και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων των αναγκών της για την ασφάλεια. Οπότε μια ε, ισχυρή έκκληση ανεξάρτητη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών υπέρ του αφοπλισμού θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διάσκεψη επανεξέτασης της συνθήκης TNP. Και μάλιστα η διάσκεψη αυτή, η ε, αξιολόγηση επανεξέτασης ε, της συνθήκης περί διάδοσης αποτελεί κοινή συλλογική ευθύνη και ανέκαθεν ε, επισημένα με την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουν δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν από το μεγαλύτερο, ε, μάλλον οι δύο πυρηνικές δυνάμεις που έχουν το μεγαλύτερο πυρηνικό προστάσιο, αλλά υπάρχει κοινή ευθύνη και συλλογή και των άλλων πυρηνικών δυνάμεων και γι' αυτό προσβλέπουμε στον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διευκολυνθεί ένα αίσιο πέρας μια θετική έκβαση της διάσκεψης του Μαΐου. Και πέραν τώρα της διάσκεψης αυτής για την επανεξέταση της συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών. Θα πρέπει να είμαστε οραματιστές και δεδομένων των αλλαγών στο περιβάλλον ασφάλειας παγκοσμίω, είναι σημαντικό να εμ, ατενίσουμε και το μέλλον μετά τη διάσκεψη του 2020. Ε, τα νέα γεγονότα και κάποιες ρηξικέλευθε εξελίξεις όπως η τεχνολογική επανάσταση καταδεικνύουν όλο και σαφέστερα ότι η παρούσα νοοτροπία περί εφοπλισμού και ο τρόπος σκέψης μας που είναι απόρρια κυρίως του ψυχρού πολέμου και της εποχής αμέσως μετά το ψυχρό πολέμου όλος αυτός ο τρόπος σκέψης θα πρέπει να επανεξαλογηθεί και να αναθεωρηθεί. Η αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας η δημιουργία ενός πολυπολικού τοπίου διεθνώς, αλλά και οι προκλήσεις και οι ε, ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες, γιατί μιλούμε πολύ συχνά για προκλήσεις, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι οι νέες τεχνολογίες επιφέρουν και νέες ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τους τρόπους ελέγχου, επαλήθευσης. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ε, συνάντησα πολλούς εμπειρογνώμονες από χώρε και ζητώ να διαμορφώσουμε ένα νέο όραμα στο μέλλον για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Και πολύ συχνά ακούω σχεδόν από όλα τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χρειάζεται ένα τέτοιο νέο όραμα. Και ένα τέτοιο νέο όραμα δεν θα πρέπει να απορρίψει το ηχερίδιο κανόνα που έχουμε σήμερα. Το μήνυμα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν σαφέ και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέως το ίδιο. Ας προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε, να προστατεύσουμε, να διατηρήσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία που έχουμε και που μας επέτρεψαν να κρατήσουμε ασφάλεια και ειρήνη στον κόσμο, να τα προστατεύσουμε και να τα διαφυλάξουμε όλα αυτά, αλλά όλοι έχουμε επίγνωση ότι οι επικοδομητικές ε, συζητήσεις ε, για τη νέα προσέγγιση για τον έλεγχο των όπλων θα είναι χρονοβόρες διαδικασίες και ταυτόχρονα θα πρέπει ε, να κάνουμε τα δύνατα δυνατά και να μην φυστούμε προσπαθειών για να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα μας, αλλά από τη σκοπιά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πολλές από τις βασικές αρχές που μας εξυπηρέτησαν μέχρι στιγμή, θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση τη παγκόσμια προσέγγιση για τον αφοπλισμό. Και δύο από αυτέ τι αρχές είναι οι πιο σημαντικέ. Η μία αφορά την απόλυτη ε, εξάλληψη των πυρηνικών όπλων και η διατήρηση του καρόνα κατά τη χρήση των πυρηνικών. Αυτέ οι δύο αρχέ θα πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν ύψιστε προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών και τη παγκόσμια κοινότητα. Γιατί είναι κοινό μα στόχο ένα κόσμο χωρί πυρηνικά. Και αυτό το στόχο θα πρέπει να τον διατηρήσουμε. Το δεύτερο είναι το εξή. Εάν θέλουμε να έχουμε τεχνολογική προσέγγιση ε, της, ε, του αφοπλισμού, ε, θα πρέπει να έχουμε την αρχή της δυνατότητας επιβεβαίωσης. Άρα όχι μόνο να συζητούμε, αλλά να μπορεί να γίνει και επιβεβαίωση. Το δεύτερο στοιχείο θα είναι η διαφάνεια και το τρίτο στοιχείο θα είναι η αρχή της μη μεταστροφής. Στην διαφάνεια ενέχονται και οι ιδέες της ε, ε, διαδικασίας ε, αναφοράς, πρέπει δηλαδή να είμαστε υπόλογοι και να μπορούμε να αιτιολογήσουμε. Είναι θεία στοιχεία τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερως, άσχετα από οποιαδήποτε επιλογή εν τέλει κάνουμε και που θα είναι κατάλληλη για τον 21ο αιώνα. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις, τα, τα στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο καλύτερα θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Θα δώσω κάποια παραδείγματα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τη νέα προσέγγιση ε, του αφοπλισμού. Ας πούμε, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα, ε, όλα τα πυρηνικά όπλα, ε, τον τρόπο παράδοσής τους, γιατί μέχρι τώρα ο αφοπλισμός αφορούσε κυρίως τον αριθμό των οπλοστασίων. Ωστόσο, πιστεύω ότι τώρα πλέον θα πρέπει να δούμε και ποιοτικά στοιχεία αυτού του οπλοστασίου. Δεν χρειάζεται να σας το πω, ωστόσο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε τον κανόνα κατά των ε, χημικών ε, όπλων ε, και οποιονδήποτε όπλων μαζικής καταστροφής που θα πρέπει να απαγορευτούν τον 21ο αιώνα. Και βεβαίως η λογοδοσία για τη χρήση τους θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πολύ σημαντική παραμένει είναι η προτεραιότητα για τα Ηνωμένα Έθνη. Ο κανόνας κατά της χρήσης των βιολογικών όπλων επίσης, καθώς επίσης και ένα πλαίσιο συντονισμένης ε, ανταπόκρισης σε περίπτωση τέτοιας χρήσης και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, θα πρέπει να δούμε και το θέμα των ε, πυράβλων γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά ε, την προστασία των ε, πολιτών, των, του αμάχου πληθυσμού θέμα, ιδιαίτερα σημαντικό ε, στην Μέση Ανατολή. Εδώ δεν υπάρχουν πραγματικά διεθνή στάνταρτ πρότυπα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πλέον. Έφτασε η ώρα να τα αντιμετωπίσουμε. Ε, η δικιά μου συμβουλή είναι ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και το σύστημα ε, της αντιπυραυλικής ε, άμυνας ε, βεβαίως πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, ωστόσο ο φόβος για αυτά τα συστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αναφέρθηκα ήδη ε, στο, στην περιφερειακή διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την περιφερειακή προσέγγιση ε, του αφοπλισμού, πράγμα που προϋποθέτει καλύτερη οικοδόμηση των μέτρων εμπιστοσύνης και προϋποθέτει επίσης ότι ο αφοπλισμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια και των πολιτικών διαπραγματεύσεων και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων επίλυσης ε, ε, συγκρούσεων και όχι μονάχα να λυθεί ε, σε επίπεδο τεχνικό, τεχνολογικό. Η διαφάνεια για τα νέα οπλικά συστήματα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια ακριβώς της ανάπτυξης νέων τέτοιων τεχνολογιών. Εξίσου όμως και μια και τα Ηνωμένα Έθνη ιδιαίτερως ασχολούνται με τα θέματα της αναπτυγμένης προστασίας των ε, πολιτών ε, θα πρέπει να δούμε και από αυτή την πλευρά. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας, κυρίως οτιδήποτε αφορά τον κυβερνοχώρο και την ε, τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να ξεχνάμε και άλλα θέματα όπως είναι οι 3D εκτυπωτές και άλλα στοιχεία τεχνολογικής εξέλιξης αναγνώριση και αντιμετώπιση επίσης ε, θεμάτων που σχετίζονται με τον αντίκτυπο των οπλικών συστημάτων και των όπλων ε, στα ε, φύλλα. Δηλαδή είναι διαφορετική, ο αντίκ, διαφορετικός ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν κάποια συστήματα σε άνδρες ή σε γυναίκες, σε αγόρια ή σε κορίτσια. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε καλύτερα τα ζητήματα αυτά. Εν τέλει, οφείλω να υπογραμμίσω πάντα από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών ότι θεωρούμε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει την ανάγκη και τη σημασία πολυεθνικών ε, λύσεων είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συμφωνίες φυσικά, αλλά ε, ε, είναι σημαντικό δηλαδή να υπάρχουν διεθνικές συμφωνίες, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και πολυμερείς ε, συμφωνίες όσον αφορά τα θέματα αυτά, εξού και ο ρόλος που μπορούν να παίξουν τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά δε την διάσκεψη της ε, συνθήκης για τη μη διάδοση, τα Ηνωμένα Έθνη θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την δύναμη πυθούς που έχουν έτσι ώστε ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι πυρηνικές χώρες και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι να συζητήσουν σε βάθος όλα τα ζητήματα ε, αυτά. Πρόκειται για κάτι το οποίο ε, θέλουμε να μελετήσουμε έτσι ώστε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ο καλύτερος χρόνος για αυτές τις διαδικασίες καθώς και τι μορφή θα πάρουν. τέλο, ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεμονωμένων κρατών μελών, καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ημών δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της ήδη παίζουν ε, σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κοινότητα του αφοπλισμού. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερως υποστηρίζει την εργασία των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα αυτών ε, και μεταξύ άλλων και με οικονομικό τρόπο αναφέρθηκα προηγουμένως στην πολιτική υποστήριξη, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ε, και την οικονομική υποστήριξη που ήταν πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά δε τις εργασίες οι οποίες οδηγούν ή στην ε, διάσκεψη αναθεώρησης ε, της συνθήκης NPT ε, που ανέφερα και προηγουμένως. Σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας και τα μικρά όπλα, μικρού βελενικού στη Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θέλουμε οπωσδήποτε να σιγουρευτούμε ότι οπωσδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιμετωπίζεται καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει σε αυτό αυτό, καθώς επίσης και όσον αφορά την μη διάδοση ε, ε, ε, των όπλων μαζικής καταστροφής σε χώρες οι οποίες δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά Ξέρετε ότι έχουμε και κάποιες νέες διαδικασίες ε, στα ε, Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε σχέδια για την μείωση της χρήσης ε, ηλεκτρικής ενέργειας, να σταματάμε τις συνεδριάσεις μας στις 6 το απόγευμα κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Μαζί με τα κράτη-μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υψώσει σημαντικά τη φωνή της από πολιτικής απόψεως στις διαπραγματεύσεις για θέματα αφοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, σημαντικές συνεδριάσεις συζητήσεις ε, στα πλαίσια του NPT και ε, συζητήσεις για άλλες πανεμφερείς ε, συνθήκες οι πολίτες επίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολύ συχνά ε, ασχολούνται άμεσα με τα θέματα των μέτρων που απορρέουν από την συνθήκη για την μη διάδοση ε, και για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και είναι σημαντικό στις διάφορες πλατφόρμες να είναι ισχυρή η φωνή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και παίζουν σημαντικό ρόλο μέσω δικών τους πρωτοβουλειών υπέρ ε, ε, του εφοπλισμού, όπως ας πούμε ε, είναι η ομάδα της Στοκχόλμης. Επίσης, ο, προ, η, πρωτοβουλία διαλόγου για τους πυράβλους στη Γερμανία, πολύ σημαντική διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και θα προχωρήσουν και οι συζητήσεις για θέματα τα οποία έχουν λίγο μείνει πίσω όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Τα ευρωπαϊκά κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης δρούν δια του παραδείγματος ε, όσον αφορά την, ε, τις δεσμεύσεις καθώς επίσης ε, και την υλοποίηση δεσμευτικών αποφάσεων. Είμαστε ευγνώμονες γιατί εσείς λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη σας τα μέτρα αυτά. Έχω σημειώσει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον αφοπλισμό από πλευράς του Κοινοβουλίου, των Κοινοβουλίων συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χάρηκα πάρα πολύ που τον προηγούμενο Οκτώβριο θα σας υποδέχθηκα ε, στα Ηνωμένα Έθνη και πραγματικά κάτι που με εντυπωσίασε ήταν ε, ότι οι συζητήσεις μας ήταν πραγματικά συζητήσεις ουσίας. Δεν ήταν ε, απλώς μια πολιτική κίνηση. είδα ότι πραγματικά σας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα ζητήματα και το ενδιαφέρον σας πραγματικά είμαστε ευγνώμονες μάλλον για το ενδιαφέρον σας. Επίσης υπάρχουν ε, εθνικά κοινοβούλια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα οποία με επισκέφθηκαν και με τα οποία είχα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Επομένως, δεν μας εκπλήσει το ενδιαφέρον Πιστεύω ότι αυτό απορρέει και από ε, τους εκλογείς σας, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, γιατί κατανοούν ότι πρόκειται για θέματα ασφάλειας δικής τους επίσης. Θα θέλαμε βεβαίως να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας ε, για, με σκοπό και στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση αυτών των συζητήσεων. Ε, θα έχουμε βέβαια και σε λίγους μήνες την ευκαιρία άμεσα να το κάνουμε αυτό, αλλά και πέρα από αυτό ε, πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τα μέλη του Κοινοβουλίου, γιατί μέσα από αυτές τις συζητήσεις, μέσα από τέτοιου είδους ε, διαλόγους, εγώ ε, παίρνω πολύ, πολλές ενδιαφέρουσες ε, ιδέες, τις οποίες μεταφέρω μετά σε άλλες περιφέρειες και τις οποίες δουλεύω και εγώ η ίδια στο μυαλό μου. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο, θα σταματήσω εδώ. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την ανταλλαγή των απόψεών μας εδώ ή αλλού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στην κυρία Τζάκι Τζόουνς, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας με τα Ηνωμένα Έθνη και μετά θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας που συνέδεσε σε αυτήν την συνεδρίαση την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις ΕΠΑ και βεβαίως ε, την κυρία Νακαμίτσου που μας ε, έκανε ε, μια πολύ μεγάλη επισκόπηση για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα ως ε, ε, πολίτες θα πρέπει να ξέρετε ότι εφόσον ε, η Βρετανία φεύγει στο τέλος της εβδομάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας ανησυχούν πολύ όλα αυτά τα ζητήματα στην Βρετανία. Δεν είναι εύκολο το έργο σας και δυστυχώς η κατάσταση παγκοσμίω δεν δίνει μεγάλη αισιοδοξία όσον αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε πολλά μέρη του κόσμου. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε βέβαιοι πως η ΟΗΕ δεν είναι μόνο σε αυτές τις προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τις αρχές της ε, και τα συμφέροντά της που είναι πολύ ευθυγραμμισμένα με τη δική σας εντολή. Θα μείνουμε ενωμένοι και θα στηρίξουμε τις εξής θέσεις. Ο μηχανισμός ε, ε, για το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και για την ε, επίλυση των διαφορών συζητήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία και με στόχο να βρεθούν λύσεις όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει προσιλωμένη στην GCPOA για, ώστε να βρούμε κοινού στόχους καθώς είναι το μόνο βιώσιμο μέσο που έχουμε για να προωθήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ε, περιοχή. Λυπούμεθα που η ΕΕ και η Ρωσία έχουν αποχωρήσει από την ε, INF, τη συνθήκη για τα πυρηνικά μέσου ελληνικούς και τους καλούμε πραγματικά να λειτουργήσουν και να δράσουν υπεύθυνα με στόχο τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσθέσει και ε, ε, τα ατού της στην απαλή δύναμη ώστε πραγματικά να μπορέσει να πείσει πυρηνικά κράτη στο να, ε, να μην επενδύουν πλέον στην περαιτέρω ανάπτυξη των οπλοστασίων τους και ε, για να πείσει χώρες που δεν έχουν υπογράψει αυτήν την συνθήκη ώστε να το πράξουν. Πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε με τη φωτιά. Η κίνδυνη είναι τεράστια. Εσείς αναφέρατε ορισμένους εξ αυτών, αλλά θέλω να αναφέρω και τα drone, τα μη επανδρομένα υπτάμενα ε, οχήματα. Επίσης ε, θέλουμε να στηρίξουμε την, ε, τον οργανισμό για τη συνθήκη της ε, ολοκληρωμένης πάυσης των πυρηνικών, εξάλληψης των πυρηνικών δοκιμών. Συμφωνούμε μαζί σας γιατί πρέπει να προστατευτούν και οι άμαχοι γιατί φυσικά είναι οι πιο ευάλωτοι σε κάθε σύραξη και αν δεν έχουμε και μελέτη όσον αφορά τον αντίκτυπο και ως προς το φύλλο ε, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άμαχους ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα τους ακούσουμε όλους και μετά θα σας δώσω το λόγο. Κινάμε με τον Σβέν Μίξερ που είναι και ο εισηγητής, όπως σας είπα της ε, έκθεσης πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Βοηθέα του Γενικού Γραμματέα Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπουμε μετά την ε, επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας μας στη Νέα Υόρκη και τη συνάντησή μας εκεί. Έχω μερικά σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της ήταν ανέκαθεν δεσμευμένα υπέρ της, του αφοπλισμού για προφανείς λόγους. Ε, γιατί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η Ευρωπαϊκή ε, η Ευρώπη ήταν το πιο πιθανό θέατρο ε, εχθροπραξιών μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων. Και όπως είπατε έχουμε και δύο από τις πέντε πυρηνικές δυνάμεις στην συνθήκη. Σε λίγο μία θα ε, εγκαταλείψει. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε συμμαχίες που δρούν βάσει συνένεσης. Και ελπίζω κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε εφοπλισμό, αλλά όσοι υπάρχουν ε, διαμάχες στον κόσμο θα εξακολουθεί η συμμαχία μας να έχει και πυρηνικά όπλα. Ένας από τους συνομιλητές μας την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι ε, είναι σχετική η πιθανή επιτυχία ή αποτυχία της διάσκεψης επανεξέτασης της συνθήκης. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια δεν καταλήξαμε σε ουσιαστικές διακηρύξεις από τις διασκέψεις ε, ε, της επανεξέτασης. Αλλά ακόμη και δεν υπάρχει τέτοια συνενετική διακήρυξη, περιστρέφεται γύρω από ελάχιστους κοινούς παρανομαστές. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν, ε, ποιος ήταν ο ορισμός της πολιτικής επιτυχίας μιας τέτοιας διάσκεψης. Η πολιτική συμφωνία γύρω από ένα συνενετικό έγγραφο είναι θεωρητικά ε, επιτυχία. Σε ό,τι αφορά την ε, ουσιαστική όμως έκβαση, τι θα θεωρούσατε εσείς επιτυχή έκβαση της ε, διάσκεψης. Επίσης, μιλήσατε για τις νέες συμμετοχές. Μέχρι στιγμής μπορούν να μπουν στην συνθήκη περί διάδοσης μόνο χώρες που δεν είναι πυρηνικές δυνάμεις. Τι θα γίνει όμως στο μέλλον. Γιατί αν σκεφτούμε κάποιες καταστάσεις ή κάποια περιστατικά όπου βρεθήκαμε στο χείλος πυρηνικού πολέμου, το 2002 για παράδειγμα, ε, τη διαμάχη Ινδίας και Πακιστάν για το Κασμίρ. Ε, εκεί φάνηκαν οι προκλήσεις που δημιουργεί η μη διάδοση. Και γι' αυτό δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Κορέα ως πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις ε, αιτήσει συμμετοχής στο, στο NPT και πώς θα προωθήσουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της συνθήκης ε, της μη διάδοσης. Επίσης, είπατε ότι μετά τη διάσκεψη επανεξέτασης θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, όπως τα αντιπυραυλικά συστήματα. Μιλήσαμε επίσης για την ε, κατάρρευση, τη λυπηρή κατάρρευση τη συνθήκης για τα πυρηνικά μεσουβεληνικούς και την ε, αποχώρηση των Αμερικανών πρώτα και μετά την διακοπή της ε, συνθήκης. αλλά οι Ρώσοι από τη συστήματα που βάσει τη συνθήκη θα ήταν απαγορευμένα. Στο μεταξύ έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο και νέοι παίκτε που δεν δεσμεύονται από αυτή οι άλλε διμερείς συνθήκε, οπότε υπάρχει ανάγκη πολυμερού συνάντηση και συνεννόησης. Ε, σε ό,τι αφορά τη, τα αντιβαλιστικά συστήματα, μήπως θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε τη συνθήκη IBM ή σκεφτόσαστε κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει δυνατότητα η συμφωνία αυτή να λάβει πιο πολυμερή χαρακτήρα, η συμφωνία δηλαδή για τα αντιπυραυλικά βαλιστικά συστήματα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ΕΛΚ τώρα, ο κύριος Κρίς Πέτερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νακάμιτσου που ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα την ευκαιρία να σας συναντήσω και στα πλαίσια της αποστολής μας στη Νέα Υόρκη και βλέπω εδώ τις σημειώσεις που είχα από τον περασμένο Οκτώβριο. Εσείς επανειλημμένως επισημάνατε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδειχθεί ως σημαντικός εταίρος στις συζητήσεις για τον αφοπλισμό. Ελπίζω με, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη να είμαστε αυτός ο ισχυρός εταίρος και να διευκολύνουμε την επίτευξη αποτελεσμάτων. Αυτό θα ήταν το πρώτο ζητούμενο και μέλημά μα. Δεύτερον, όπως αναφέρατε, για τα Ηνωμένα Έθνη είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Γενικός Γραμματέας έχει το δικό του πρόγραμμα ε, για τον αφοπλισμό και το προβάλλει και έχει τον αφοπλισμό ως προτεραιότητα και πιστεύω ότι σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα μπορούμε να βρούμε λύσεις ε, και με άλλους εταίρους. Επίσης στη Νέα Υόρκη μας είχατε πει ότι χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα και μια νέα προσέγγιση και εδώ μας είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη, τις κυβερνοπηλές και άλλα στοιχεία. Είπατε όμως ότι χρειαζόμαστε και εμπειρογνωσία. Έχουμε ανάγκη από εμπειρογνώμονες για να μας ε, ε, ενημερώσουν για τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες αυτές ρηξικέλευτες τεχνολογίες και τι κινδύνους εμπεριέχουν. Τι γίνεται τώρα αυτήν την ανάγκη εμπειρογνωσίας, την ανάγκη συζήτηση με εμπειρογνώμονες για αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνοαπειλές. Στη Νέα Υόρκη είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε πρώτα άτυπες συζητήσεις για τρία-τέσσερα χρόνια, ώστε να συγκεντρώσουμε εμπειρογνωμοσύνη και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για να διαμορφώσουμε αυτή τη νέα προσέγγιση και το νέο όραμα και να το υλοποιήσουμε. Τώρα, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ε, η Βορείου Κορέας και Ιράν, αλλά είναι πολύ σημαντικές, κυρίως όμως σχέσεις ΙΠΑ και Κίνας. Γιατί θέλουμε μια πολιτική ε, προκαθοδήγηση, ένα πολιτικό ηγετικό ρόλο για να καταλήξουμε στη συμφωνία. Υπάρχει αρκετή τέτοια πολιτική ηγεσία για να καταλήξουμε σε λύση. Δεν το βλέπω, γιατί όταν βλέπουμε τις συζητήσεις είπα και Κίνας, ε, με συμμετοχή και Ρωσίας πολλές φορές, μας προβληματίζουν οι εξελίξεις. Ναι, σίγουρα θέλουμε εμπειρογνώμονες, αλλά υπάρχει πολιτική ηγεσία, υπάρχει πολιτική καθοδήγηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρο για την αναζήτηση λύσεων, αλλά τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ηγετικό ρόλο και πολιτική βούληση για την ανέβρεση λύσεων. Για το Renew Europe, ο κύριο Φιλ Μπάνον έχει το λόγο. Με κάλυψαν οι συνάδελφοι για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ κάποια σχόλια από την κυρία Νακάμιτσου για το τι προσπάθειες έγιναν μέχρι τώρα ε, για να σε, λάβει δηλαδή, μέρος και το Πακιστάν. Ασχολήθηκα με την έκθεση για τις σχέσεις μας με το Πακιστάν και επικεντρώθηκα και στο θέμα του Κασμίρ. Πώς μπορούμε να προσετεριστούμε το Πακιστάν, τι προσπάθειες μπορούν να γίνουν για να ενταχθεί στη συνθήκη. Θα έχει κάποιο πλεονέκτημα η συμμετοχή του Πακιστάν ως συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης αν κάποια πυρηνικά προσθέσεις είναι εκτός του συστήματος, ε, ότι, διά, ότι μέγεθος και να έχουν, ίσως ε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και είχα και μια ερώτηση για το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, αλλά απαντήθηκε η απόρρια μου. Για το ΕΛΚΟ, κύριος Μπασέσκου. I, I have a observation. Έχω μια παρατήρηση. Όλοι εμείς μιλάμε για τη Ρωσία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν κάνουμε λόγο για την συμφωνία INF ή όταν ε, λέμε ότι θα πρέπει να μειωθούν τα πυρηνικά οπλιστάσια κλπ. Κατά την γνώμη μου όμως και λαμβάνοντας υπόψη την ε, εμπειρία μου, εγώ καταλαβαίνω κάποιες σημαντικότατες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ρωσική Ομοσπονδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπόθεση ότι η Κίνα μένει έξω από αυτές τις συμφωνίες και αυτή τη στιγμή και οι δύο, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ρωσική Ομοσπονδία, βλέπουν εν τέλει ότι απέναντί τους έχουν την Κίνα με ένα οπλοστάσιο σχεδόν ε, ίδιο με το πυρηνικό οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, και λαμβάνοντας υπόψη τούτη την κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να ζητούμε σεβασμό από πλευράς Ρωσίας και ΙΠΑ των αποφάσεων. Μόνο οι πολυμερείς ε, αποφασίσεις είναι αυτές και δεσμεύσεις είναι αυτές οι οποίες θα επιτρέψουν την πρόθεση των διαπραγματεύσεων και θα διασφαλίσουν την τελική επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, When... πώς μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές τις πέντε μεγάλες χώρες εάν δεν λύσουμε το πρόβλημα των δευτερογενών παικτών όπως Βόρεια Κορέα, Ιράν, Πακιστάν, ε, Ινδία. Από στρατηγικής απόψεως τα ε, ε, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να έχουν όλα τα, όλα τα κράτη αυτά την ιδέα να ασκήσουν πίεση ε, στις χώρες αυτές οι οποίες θα πρέπει να δεχτούν να καταστρέψουν το πυρηνικό τους ε, οπλοστάσιο. Και μετά τα μόνιμα μέλη θα πάρουν μια απόφαση. Βέβαια ακόμα είμαστε πολύ μακριά από τη στιγμή που ε, θα πάψει να υπάρχει πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο τούτο. Ίσως καλύτερο θα ήταν να προσδοκούμε ε, μια μετριοπαθή ας πούμε επιτυχία στην επόμενη αναθεωρητική διάσκεψη και να προσπαθήσουμε περισσότερο να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους ε, δευτερογενείς παίκτες και εκεί να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Κοιτάξτε, εσείς ε, συγχαίρετε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει σε αυτήν την πολιτική προσπάθεια του αφοπλισμού ή και την προσπάθεια ε, ολικής κατάργησης των πυρηνικών. Ναι, θα πρέπει να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λιγότερη δυνατότητα επιρροής ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα όλο και περισσότερο χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη στρατιωτική δύναμη και πολλές στρατιωτικές και πολλούς στρατιωτικούς πόρους ε, στην ουσία δρούν χωρίς να σέβονται την διεθνή ε, τάξη ε, προσπαθώντας να επιβάλλουν κάποιες λύσεις. Ή πρόκειται για περιφερειακές λύσεις, λύσεις δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο, δόξα τω Θεώ. δεν έχουν γίνει ακόμα παγκόσμιες λύσεις. Ε, ωστόσο έχουμε την Λιβύη, ας πούμε, τους τελευταίες ε, εβδομάδες έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες υπαγόρευσαν στην ουσία τις κινήσεις και σε αυτή την περίπτωση η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν μεγάλη και δεν διατηρήθηκε περιπτώσει. Σε πραγματικούς όρους ε, επανειλημμένα στην Επιτροπή μας έχουμε γύρει ε, τα σχετικά ζητήματα. Και τι σημαίνει μια Ευρώπη χωρίς στρατιωτικές ε, δυνάμεις και πόσο μπορεί μια τέτοια Ευρώπη να επηρεάσει όποιες αποφάσεις. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις από τη δική μου πλευρά σε σχέση με τα όσα μας είπατε. Ένα συμπεράσματι εγώ λέω ότι μονάχα μέσα σε ένα κλίμα πολυμέρειας και σε αντίληψη πολυμέρειας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί διαφορετικά ουδόλως βλέπω δυνατότητα λύσης. Και δεν τα βλέπω, εν πάση περιπτώσει, καθόλου καλά τα πράγματα όσον αφορά μια ενδεχόμενη επιτυχία έκβαση αυτή τη αναθεωρητική διάσκεψης. Ωστόσο, σα συγχαίρω και σα εύχομαι καλή επιτυχία. Ε, ο κύριο Μπουσνέρ για του Πράσινου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Ιδίως δε όσον αφορά το τακτικό σκέλος των πυρηνικών ε, όπλων. Εδώ εγώ βλέπω να υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος όσον αφορά τη χρήση των όπλων. Ας πούμε στο Κασμίρ, όπου ε, πολύ συχνά έχει φτάσει στο πρόθυρο ε, της χρήσης τέτοιων όπλων η κατάσταση. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μιλήσαμε εδώ, έγινε λόγος για την συνθήκη με το Ιράν. Να μην λησμονούμε ότι ε, η συνθήκη αυτή δεν ανεστάλει ε, λόγω ε, συγκρούσεων. Ε, ξέρετε ότι από πλευράς των Αγιατολάχ, από πλευράς των επαναστατικών συμβουλίων της χώρας, υπάρχει ανασχετική διαδικασία. Και η γενικότερη κατάσταση σημαίνει ότι εάν κανείς προσεγγίζει τα πυρηνικά όπως το κάνει η Ευρώπη, ε, πιστεύω ότι είναι μια πολύ ασφαλμένη προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε μια συνθήκη η οποία να είναι ενδιαφέρουσα για το Ιράν και να ε, μπορέσει να την αποδεχτεί το Ιράν. Merci. Et Ευχαριστώ πολύ για το Ισιάρη κυρία Αγγιλάρ. Και θα έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν αυτό το γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση θέλω να υποβάλω μόνο. Θα ήθελα να μου πει η κυρία Νακαμίτσου ποια είναι η άποψή της ε, σε σχέση με το Ιράν ε, όσον αφορά το JCPOA και την ε, διαδικασία επίλυσης διαφορών. Αυτό ήθελα να μάθω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε πολλές ερωτήσεις κύριε Νακαμίτσου, ερωτήσεις οι οποίες ε, καταδεικνύουν ακριβώς το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο διαπιστώσατε κι εσείς άλλωστε. Και θέλω να πω στον κύριο, στην κυρία και στον κύριο Μπάνιο να τους ευχαριστήσω γιατί είναι η τελευταία ε, φορά που βρίσκονται εδώ μεταξύ τους και πραγματικά και μετά από αυτά που ε, ρώτησαν και την τοποθέτησή τους κατανοούμε ότι θα μας λείψουν πάρα πολύ. Um, these are all very difficult. Σας ευχαριστώ. Πολλές και δύσκολες ερωτήσεις. Ερωτήσεις που μας προβληματίζουν και εμάς τα Ηνωμένα Έθνη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσε περισσότερε μπορώ. Καταρχήν, το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση και μηχανισμό επίλυση των διαφορών του JCPOA. Ακούσαμε τι είπαν τα, τα τρία ευρωπαϊκά κράτη-μέλη που ενεργοποίησαν το μηχανισμό με στόχο να διαφυλάξουν αυτό το πλαίσιο και τους κοινού μας στόχους, γιατί το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το JCPOA, ήταν από τα πιο σημαντικά διπλωματικά επιτεύγματα στα θέματα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Οπότε, μακάρι οι Ιρανοί να βελτιώσουν τη συμμόρφωση του κοινού ολοκληρωμένου σχέδιου δράσης και όταν τα κράτη-μέλη εξηγούν ότι προσπαθούν να ετοιμάσουν για αυτό το λόγο ε, μια πλατφόρμα για να έχουν διάλογο με τους Ιρανούς και να επιλύσουν τις διαφορές, το χαιρετίζουμε. Εμείς στη γραμματεία του ΟΗΕ δεν έχουμε επίσημο ρόλο σε αυτό το μηχανισμό επίλυσης των διαφορών και επί του παρόντος απλώς παρακολουθούμε προσεκτικά τη διαδικασία και ουσιαστικά λέμε το ίδιο με τα τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να διαφυλάξουμε τη συμφωνία αυτή και το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Και αν θεωρούν τα μέρη ότι μπορούν και τα Ηνωμένα Έθνη να παίξουν κάποιο ρόλο, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Εν τω μεταξύ πάντως δεν έχουμε κάποιον επίσημο ρόλο. Πάντως συμμεριζόμαστε τον στόχο της ε, διαφύλαξης της συμφωνίας και της επίλυσης της διαφοράς. Για το New Start, τη νέα συμφωνία για τη μείωση στρατηγικών όπλων. Συμφωνώ απόλυτα και ακούσαμε επανειλημμένως και το Γενικό Γραμματέα αλλά και την υποφαινόμενη να κάνουν δηλώσει προ αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμε ε, ζητήσαμε επανειλημμένως και επισταμένως την παράταση αυτής της συμφωνίας, της νέας συμφωνίας για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, ε, που αν γίνει μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο θα είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις δεν θα έχουν πια κανένα περιορισμό για το προστάσιό τους αν δεν παραταθεί η συμφωνία αυτή του χρόνου και αυτό θα είναι πολύ επικίνδυνο για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση προς τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη να συμφωνήσουν και να επεκτείνουν, να παρατείνουν αυτή τη νέα συμφωνία. CTBT, Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Πρόκειται για μια αμυγή συμφωνία αφοπλισμού που την περιμέναμε φυσικά, έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ και όσο το συντομότερο τεθεί σε ισχύ τόσο το καλύτερο και μάλιστα όλοι και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες χώρες, όλες οι χώρες που υπέγραψαν την συνθήκη αυτή. Αυτό ζητούν επανειλημμένως ε, και κάθε χρόνο στα Ηνωμένα Έθνη μετεπιτάσεως. Συνήθως γίνονται διασκέψεις υψηλού επίπεδου, σε επίπεδο υπουργών κυρίως για τη συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπλοκη κατάσταση, συμφωνώ απόλυτα. Και όταν λέμε θεμητές ε, ανησυχίες περί ασφάλειας, αυτό εννοούμε. Οι θέσεις είναι διαφορετικές και περίπλοκες ανάλογα με τα συμφέροντα κάποιας χώρας, με την ε, γεωγραφική της θέση και τις συμμαχίες τις οποίες συμμετέχει. Και το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μας για μια επικοδομητική συζήτηση στην αναθεωρητική διάσκεψη της συνθήκης μη διάδοσης και γενικώ για οποιαδήποτε συζήτηση περί εφοπλισμού και ελέγχου των όπλων είναι να αντιληφθούμε τις εύλογες και θεμητές ανησυχίες για την ασφάλεια που έχουν όλα τα κράτη-μέλη και να δείξουμε κατανόηση για αυτές. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούμε, συνέβη αυτό στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε για αυτό το θέμα, ότι μερικές φορές τα συμβαλόμενα κράτη υιοθετούν ε, μια περιτά εχθρική στάση στη συζήτηση. Και μια τέτοια αρνητική συμπεριφορά σίγουρα δεν βοηθά τα κράτη για μια γνήσια και ουσιαστική συζήτηση επί τη βάση των θεμητών ανησυχιών όλων των μερών. Πιστεύω ότι είναι η ώρα να επιστρέψουμε σε μια πολιτισμένη συζήτηση όπως ζητούν ε, πολλά κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη που το διατείνονται είναι και τα πιο θαραλέα και υπενθυμίζουν στους ομολόγους τους ότι οι συζητήσει είναι πολύ σημαντικέ και δεν θα πρέπει να τις ε, τορπιλήσουμε, να τις υπονομεύσουμε πριν περάσουμε στην ουσία της συζήτησης. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι οι θέσει των ε, κρατών μελών είναι πολύ περίπλοκες. Και τι θα θεωρούσα επιτυχία. Αυτό μονίμως είναι ένα μπαλάκι που το επιστρέφω στα συμβαλόμενα κράτη της συνθήκης. Ε, πολλοί λένε μία φιλόδοξη έκβαση ε, και πολυσχηδή σαν αυτή του 2010 μάλλον δεν είναι ρεαλιστική προσμονή και μάλλον θα συμφωνούσα ότι το σημερινό περιβάλλον δεν είναι πρόσφορο για μία ε, γενική και φιλόδοξη ε, συνενετική διακήρυξη ως αποτέλεσμα της διάσκεψης. Και εδώ και 1,5 χρόνο ζητώ από τα συμβαλόμενα κράτη της συνθήκης να προσδιορίσουν ή να καταλήξουν σε μια κοινή αντίληψη για το τι θα θεωρούσαν επιτυχή έκβαση της αναθεωρητικής διάσκεψης. Και αν προσδιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας και ξέρουμε ποιο είναι το απαραίτητος ελάχιστο επίτευγμα, θα μπορούσαμε σε αυτή την ψαλίδα να καταλήξουμε σε ένα κοινό όραμα για το δυναμικό της έκβασης της διάσκεψης περί επανεξέτασης. Και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε και τις συγκεκριμένες συζητήσεις, ακόμη και για ε, το, τη μορφή της έκβασης. Δεν υπάρχει κάτι στερεότυπο, δεν έχουμε κάποια στερεότυπη διακήρυξη. Το έγγραφο του 2020 θα είναι γενικό και περιεκτικό, αλλά δεν υπάρχει κανένας απαράβατος κανόνας ότι θα πρέπει το τελικό έγγραφο να έχει σώνει και καλά συγκεκριμένη μορφή. Οπότε τα συμβαλόμενα κράτη θα πρέπει να ανασκουμποθούν και να περάσουν στη δουλειά. Και περιμένω με ανυπομονησία την αυριανή μου συνάντηση στη Γενέβη και με τον οριθέντα πρόεδρο της διάσκεψης, γιατί Πραγματικά αυτό θα συντονίσει τι συζητήσει με τα συμβαλόμενα κράτη και θα προσπαθήσει από κοινού μαζί του να διαμορφώσει ένα κοινό όραμα για την επιτυχή, την αίσια έκβαση τη διάσκεψη. Και ποιο θα ήταν το απολύτω απαραίτητο αποτέλεσμα, το ελάχιστο απαραίτητο αποτέλεσμα, αλλά και τη μορφή του τελικού εγγράφου, εγγράφου ή εγγραφών της διάσκεψης. Το θέμα Ινδίας και Πακιστάν όντως ε, ακαθόδες ε, και δυσεπίλητο αυτό το θέμα και οι χώρες που είναι πυρηνικές δυνάμεις και βρίσκονται εκτός του πλαισίου της συνθήκης περί ε, είναι δύσκολο ζήτημα. Γιατί οι πέντε πυρηνικές δυνάμεις εντάσσονται στο πλαίσιο του TMP οι συνθήκε περί μη διάδοση των πυρηνικών. Όσοι βρίσκονται εκτό αυτού του πλαισίου και επειδή δεν υπάρχει ακόμη πολυμερή πλατφόρμα που να λειτουργεί και σίγουρα η διάσκεψη για, την, για τον αφοπλισμό αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε, αλλά εδώ και 20 χρόνια και δεν είχαμε ουσιώδει συζητήσει και διαπραγματεύσει για τον αφοπλισμό. Οπότε δεν έχουμε μια πραγματικά εύρυθμη και λειτουργούσα πλατφόρμα, πολυμερή πλατφόρμα για τα θέματα αυτά. Οπότε μετά από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες και συζητήσεις που κάναμε, ένα από τα στοιχεία που εντόπισα είναι ότι ίσως χρειάζονται πιο περιφερειακές προσεγγίσεις. Και εννοούσα ακριβώς και αυτά τα θέματα. Θέματα όπως ε, διαφορά Ινδίας και Πακιστάν. Αν δεν λύσουμε ή δεν κατευνάσουμε τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο αυτών χωρών, δεν μπορούμε να έχουμε συζητήσεις περί εφοπλισμού. Το θέμα δεν είναι τεχνικό που θα πρέπει να εξεταστεί μόνο ως τεχνικό θέμα εφοπλισμού, αλλά εντάσσεται στη γενική συζήτηση για την πολιτική ασφαλείας. Πάντως, μία από τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που είχαμε ήταν η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, που πρόσφατα, πέρυσι συγκεκριμένα, εγγενίασε τη διαδικασία της δημιουργίας κλίματος πρόσφορου για, την για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Ήταν πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Και μάλιστα συμπεριέλαβαν στις συζητήσεις και την Ινδία και το Πακιστάν. Χτύπησαν όλες τις κατάλληλες πόρτες για τον πυρηνικό διάλογο. Και βέβαια είναι μια διαδικασία διαλόγου, αλλά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πιστεύω ότι θα φέρουν κοντά και πυρηνικές δυνάμεις του, της συνθήκης και πυρηνικές δυνάμεις που είναι εκτός του πλαίσιου της συνθήκης και αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και είναι από τα πιο ε, δύσκολα και τα πιο σημαντικά θέματα αν είμαστε πραγματικά σοβαροί για την, για την εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Αμφιβάλλω όμως αν οι χώρες ε, που είναι πυρηνικές δυνάμεις ε, που είναι εκτός του TMP θα μπορούσαν να προσχωρήσουν ως μη πυρηνικές ή αν θα γίνουν κάποιες προσαρμογές, αλλά πολύ αφιβάλλω. Σε ό,τι αφορά τα α, αντιπυραυλικά συστήματα, βαλιστικά αντιπυραυλικά συστήματα, δεν έχω κάποια παγιωμένη α, άποψη, όπως και για τα γενικά αντιπυραυλικά συστήματα. Το θέμα αυτό των αντιβαλιστικών πυράβλων είναι τα πιο ευαίσθητα και σημαντικά. Και αν ε, δεν συζητήσουμε αυτά τα συστήματα αντιβαλιστικών πυράβλων με τα γενικά συστήματα παράδοσης πυράβλων, αν δεν τα συζητήσουμε αυτά από κοινού, πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το, τον έλεγχο των όπλων και το σκοπό της του απότερου αφοπλισμού. Κοιτάξτε την περίπτωση του Ιράν. Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράση, το κοινό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράση δεν περιέλαβανε θέματα πυράβλων, γιατί ακριβώ ήταν τα πιο καθόδη και δύσκολα. Μέχρι στιγμή αυτό είναι το κενό που υπάρχει στον έλεγχο όπλων και τον αφοπλισμό, το θέμα των αντιβαλιστικών πυράβλων. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το περιλάβουμε και αυτό στι συζητήσει. Η ανάπτυξη νομοσύνης και δυνατοτήτων. Ε, εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάποια ε, πράγματα. Όσον αφορά την θέματα νέας τεχνολογίας, ναι, βεβαίως χρειαζόμαστε επιγόντως οι ηθήνοντες για τη χάραξη πολιτικής να κατανοούν καλύτερα τι συμβαίνει ως προς την τεχνολογία. Υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, Ελπίζω πως ε, όντως όσοι παρακολουθούν τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ε, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογικές επιτυχίες, αλλά ένα παράδειγμα ενός ε, μια συζήτηση πολυμερούς που κάναμε το περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο του ομάδα εργασίας για την θέματα κυβερνοασφάλειας μας ανατέθη να διοργανώσουμε πάνω από 100 συναντήσεις ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα, τον εκπαιδευτικό τομέα, ε, ε, και οι οποίοι ήρθαν στον ΟΗΕ και ε, συνεργάστηκαν και με εκπροσώπους ε, κρατών και, και των κυβερνήσεων και υπήρχε μια καλή αίσθηση ότι πραγματικά βοηθά στο να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο είναι το διακύβευμα και τι είδους τι χρειάζεται και από την πλευρά των τεχνικών ε, ε, και από την πλευρά των πολιτικών. Δημιουργούμε δηλαδή κάποιες τέτοιες πλατφόρμες δημιουργικής συζήτησης για τις κοινότητες των διπλωματών αλλά και ε, των επιχειρηματιών. Κάτι άλλο αφορά τις δυνατότητες κατάρτισης επιμόρφωσης διαφόρων κρατών μελών. Αυτό που ακούμε από πολλά κράτη-μέλη είναι ότι Στη διάρκεια του ε, μεταψυχροπολεμικής περίοδου, πολλοί ε, που ασχολούνταν με την ειρήνη και την ασφάλεια μετακινήθηκαν ε, από τον αφοπλισμό στα θέματα διατήρησης της ειρήνης. Όμως ε, καταλαβαίνουμε πως τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του αφοπλισμού και γι' αυτό πιστεύουμε πως υπάρχει ε, χώρος για, την, για τη δημιουργία δυνατοτήτων και ε, δυνατοτήτων κατάρτισης. Γι' αυτό όμως όχι μόνο για τον διπλωματικό κόσμο αλλά και για τις νεότερες γενιές ανθρώπων που ε, μπορεί να ενδιαφέρονται περισσότερο για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνεδρίαση η νεότητα υπέρ του αφοπλισμού στη Νέα Υόρκη. Ήταν άμεσο αυτό αποτέλεσμα από την πρώτη νέα εντολή της Επιτροπής που λάβαμε για να συνεργαστούμε με τους νέους. Και για πρώτη φορά θα προσφέρουμε ευκαιρίες σε νέους φοιτητές πανεπιστημίων ε, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητε μας σε αυτό το τομέα. Τώρα, θα θέλαμε ναι, να έχουμε περισσότερες επαφές με τους πολιτικούς ηγέτες. Τούτου λεχθέντος ε, γίνονται προσπάθειες Έχουμε το πλαίσιο συντονισμού P5. Ε, τελευταίος συντονιστής ήταν η Κίνα, η οποία πραγματικά προσπάθησε σε αυτό το πλαίσιο. Νέο συντονιστής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπω πως και το Ηνωμένο Βασίλειο επενδύει σε αυτήν τον συντονισμό των ΝΗ5, των 5 δηλαδή πυρηνικών κρατών και ελπίζω πως έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο ισχυρή πολιτική δήλωση από τα κράτη πέντε πυρηνικά όπλα που θα επιβεβαιώσουν την προσήλωσή τους στο άρθρο 6 της Συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών. Δεν είναι μόνο το άρθρο 6, αλλά είναι όλοι τρεις πυλώνες και θα ήταν πραγματικά σημαντικό κάτι τέτοιο, γιατί κατά τη γνώμη μου θα σχημάτιζε ένα από τα στοιχεία τα οποία θα στηρίξουν την επιτυχία ε, της συνέλευσης του Απριλίου-Μαΐου. Γίνονται τώρα πολλές συζητήσεις για το πού εντάσσεται η Κίνα και αν εντάσσεται πολύ δύσκολο θέμα, ε, το οποίο πιθανότατα θα πρέπει να το ξανααντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο πιο ειλικρινούς και γνήσιου διαλόγου ανάμεσα στα, ε, κράτη, τα πυρηνικά κράτη. Είπα πως πρόκειται για κοινή προσπάθεια, είναι όλων ευθύνη, αλλά βλέπω, εάν εξετάσουμε το 90% των ποινικών οπλοστασίων, τα, έχουν, τα κατέχουν οι δύο χώρες που ξέρουμε, δηλαδή είπα και ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα λοιπόν εκείνοι φέρουν, βρίσκονται σε μια ειδική κατηγορία ευθύνης και διαρκώς ε, ε θυμίζουμε την ιδιαίτερη ευθύνη των ε, πυρηνικών υπερδυνάμεων. Αυτό σημαίνει όμως ότι σε στον κόσμο μας, αυτές οι χώρες θα πρέπει όντως να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Όταν ε, μιλάμε με, συνομιλούμε με τους Κινέζους συνάδελφους, ε, λέω πάντα ότι το γεγονός ότι αυτά, αυτές οι εκκλήσεις προέρχονται από τις διάφορες, διάφορα μέρη του κόσμου σημαίνει αναγνώριση πως η Κίνα αυτή τη στιγμή θεωρείται υπερδύναμη και άρα φέρει αυτή την ευθύνη. Γιατί είπα όλες αυτές οι χώρες είναι εταίροι στον αφοπλισμό. Συνεργάζομαι πολύ στενά με τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Κίνα και αυτό απλά και μόνο διότι αυτές είναι οι πυρηνικές δυνάμεις οι οποίες εάν κανείς δεν κατανοεί τις θέσεις τους και ποια μπορεί να είναι τα στοιχεία που μπορεί να τις κάνουν να μετακινηθούν από αυτές τους τις θέσεις, δεν, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς και της ευθύνη του ΟΗΕ και γι' αυτό συνεργαζόμαστε ως εταίροι με αυτά τα κράτη και είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Όσον αφορά τα μικρά τακτικά πυρηνικά όπλα, ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους ε, υπογραμμίζουμε την ε, διατήρηση της αρχής της μη χρήσης ε, είναι ακριβώς ε, λόγω αυτής της νέας ορολογίας που πλέον μπαίνει στην συζήτηση και μπορεί κανείς να έχει την εντύπωση ότι είναι μικρής δύναμης αλλά εμείς δεν θέλουμε καθόλου να χρησιμοποιηθούν αυτού του είδους τα όπλα αυτά τα λεγόμενα ε, μικρά πυρηνικά όπλα είναι ε, πολύ πιο δυνατά από αυτά ε, της Χειροσύμα και του Ναγκασάκη. Και επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτά τα τακτικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκρούσεις και εμείς δεν πιστεύουμε αυτήν την ε, χρήση. Θέλουμε ε, να μην ε, να απαγορευτεί συνολικά η χρήση και να δεσμευτούν τα κράτη. Ανέφερα ήδη το Ιράν και τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ευελπιστώ αυτή είναι η ελπίδα μου ότι θα υπάρξει ευκαιρία να βρούμε λύσει σε αυτήν την ε, υφιστάμενη διαμάχη, αυτήν την διαφορά. Ε, προς ε, δεν έχουμε συγκεκριμένο επίσημο ρόλο. Εάν μπορεί να κάνουν οτιδήποτε τα Ηνωμένα Έθνη, οπωσδήποτε είμαστε έτοιμοι να σταθούμε στο ύψος του ρόλου μας. Και υπογραμμίζω για μία ακόμα φορά ότι από άποψη μη διάδοση των όπλων ή, ε, ε, το κοινό ε, συμμετοχικό σχέδιο δράσης GCPOA εξακολουθεί να ισχύει. Αυτά ήθελα να πω προσπάθησα ε, να απαντήσω στις περισσότερες τουλάχιστον από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ε, για την διαθεσιμότητα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρίβεια ε, των απαντήσεών σας. Νομίζω ότι εξ ονόματος όλων μπορώ να σας ευχηθώ καλό κουράγιο και την απόλυτη στήριξη βεβαίως να εκφράσω τη Επιτροπής μας ε, σε αυτήν την ισχυρή δέσμευσή σας. Όσον αφορά τα μέλη της Υποεπιτροπής, να σα πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα τη 17η Φεβρουαρίου ε, στις 2.30. 2.30. Ευχαριστώ.